Παρακαλώ, για να μην χάσουμε χρόνο καθόλου, θα αρχίσουμε αμέσως. Είμαστε στο σημείο 10. Χαιρετίζω εδώ την παρουσία του Μάριου Ντράγκη. Αυτή τη φορά έρχεται για να μας μιλήσει για το και για την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Συστημικών Κινδύνων και μετά από τα λίγα λόγια που θα μας πει θα γίνει η ανταλλαγή απόψεων. Σας υπενθυμίζω ότι έχει έρθει ως πρόεδρος του ΕΣΣΚ, γι' αυτό παρακαλώ να περιορίζετε τα ερωτήματά σας όταν έρθει ο καιρός των ερωτημάτων, όχι για γενικά θέματα της ΕΚΤ, αλλά ειδικά για αυτή την Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων. Σας υπενθυμίσω ότι εμείς ζητήσαμε του ζητήσαμε να έρθει και να γραφτεί χωριστά αυτή η έκθεση για το διαχωρισμό των ρόλων μεταξύ Κεντρικής Τραπέζης και Επιτροπής Συστημικών Κινδύνων. Ορίστε Μάριε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, με χαρά είμαι σήμερα ενώπιον της Επιτροπής σας να παρουσιάσω την πρώτη ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, ESRB έχετε όλοι λάβει μια, ένα αντίγραφο της έκθεσης και δημοσιοποιείται όπως μιλάω. Στις παρατηρήσεις μου σήμερα δεν θα επαναλάβω το περιεχόμενο της έκθεσης. Αντί γι' αυτό θα επικεντρωθώ σε τρεις τομείς κλειδιά της εργασίας ε, τον τελευταίο χρόνο της, του ESRB που θα μας απασχολήσουν και για το προβλέψιμο μέλλον. Αυτοί οι τρεις τομείς είναι ένα η αποτίμηση των συστημικών κινδύνων, η δημιουργία ενός υγιούς μακροπροληπτικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μεσοπρόθεσμες ε, διαφορετικές εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό σύστημα της Ένωσης. Πριν από λιγότερο ένα χρόνο το ESRB ε, προειδοποίησε ότι η κίνδυνη για το χρηματοπιστωτικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει συστημική. Μετά μια περίοδο σταθεροποίηση ε, με βάση τι ενέργειε των κεντρικών τραπεζών και άλλων ε, ιδρυμάτων νωρίτερα φέτο, πρόσφατα υπήρξαν ορισμένε εξάρσει αστάθεια και αβεβαιότητα, αλόχη του επίπεδου του Νοεμβρίου 2011 και παραμένουν θεμελιώδει προκλήσει, κατά τη γνώμη μου. Αυτέ περιλαμβάνουν την, τον περιορισμό τη ε, μετάδοση μεταξύ των κρατών μελών τη Ένωση. Δεύτερον, την προώθηση ενός, μιας μακροοικονομικής στρατηγικής που μαζί με την ε, φορολογική εξυγίανση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και θα προωθήσει τις ε, προσαρμογές ανταγωνιστικότητα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν οικονομικέ ανισότητε στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με αποφασιστικό και βιώσιμο τρόπο είναι προϋπόθεση για να επιτύχουν τα μέτρα για να υπάρξει ένα πιο ανθεκτικό χρηματοοικονομικό σύστημα που να μπορεί να μας παρέχει σε βιώσιμη βάση τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για να υποστηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα. Από μια μακροπροληπτική άποψη τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν πρώτον να εφαρμόζονται αξιόπιστοι μηχανισμοί για την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση των τραπεζών όπου χρειάζεται και την βελτίωση της επιτήρησης των τραπεζών και της επίλυσης των προβλημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο παρελθόν, το ESRB έχει υπογραμμίσει την ανάγκη όλες οι εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές να δράσουν και μάλιστα ενιαία, με ταχύτητα, φιλοδοξία και απόλυτη αποφασιστικότητα για να διασφαλίσουν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σήμερα επαναλαμβάνω αυτήν την έκκληση αναγνωρίζοντας ωστόσο τις προσπάθειες που έχουν μέχρι στιγμής γίνει. Στα πλαίσια του ευρύτερου οικονομικού και χρηματοπιστωτικού πλαισίου, το χρηματοπιστωτικό σύστημα αντιμετωπίζει ακόμη την πρόκληση προσαρμογής για να αντιμετωπίσει τις ανισορροπίες που συσσωρέθηκαν κατά το παρελθόν. Για τις τράπεζες, ήδη έχει σημειωθεί πρόοδος ε, σε διάφορα μέτωπα, αλλά χρειάζεται περισσότερη πρόοδος. Για άλλους τομείς είναι σημαντικό οι διεθνείς και ενωσιακές μεταρρυθμίσεις που έχουν στόχο να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα να εφαρμοστούν πλήρως και να γίνουν σεβαστές. Θα επανέλθω σε αυτό. Το ESRB ασχολείται με δύο πλευρές των προσαρμογών στον τραπεζικό τομέα. Πρώτα πρέπει να γίνει με συντεταγμένο τρόπο για να στηρίξει πλήρως την οικονομική ανάπτυξη χωρίς να επιδεινώνει την ευαισθησία της αγοράς και την θέση άλλων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεύτερον, ο βαθμός αναπροσαρμογής για τον ε, τραπεζικό τομέα της Ένωσης πρέπει να είναι επαρκής για να επανέλθει η εμπιστοσύνη στην φερεγγιότητα των ε, τραπεζικών ισολογισμών. Όσον αφορά το πρώτο σημείο, τα στοιχεία και έρευνα από πολλές χώρες της Ένωσης μας δείχνουν μια κάποια σταθεροποίηση των οικονομικών συνθήκων ε, κατά το πρώτο τμήμα του παρόντος έτους. Όμως οι πρόσφατες αναταράξεις υπογραμμίζουν την αβεβαιότητα που αφορούν τις προοπτικές για αυτές τις οικονομικές συνθήκες λόγω της σύνδεσής τους με την φερικιότητα των ισολογισμών των τραπεζών της Ένωσης και την άμεση και έμεση σύνδεση αυτών των ισολογισμών και την έκθεσή τους σε κρατικά ομόλογα. η στενή επιτήρηση και η συστημική αποτίμηση της ε, εφικτότητας και της φύσης των ε, προσαρμογών των τραπεζών είναι ζωτική σημασία. Το ESRB κάλεσε τους εταίρους της ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Επιτήρησης που είναι οι αρχές επιτήρησης σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο να συλλέγουν τακτικά εξάντε αναλυτικά στοιχεία από τις τράπεζες και άλλους ε, πέκτες κλειδιά του συστήματος και να τα μεταδίδουν στο ESRB. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τις τελευταίες εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στη συνάντησή του τον Ιούνιο. Να στραφώ τώρα στην εργασία που έχουμε αναλάβει για να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες του προκρισιακού πλαισίου για να, προλαμβάνουμε και να μετριάζουμε τους συστημικούς κινδύνους στην Ένωση. Το ESRB ξεκίνησε. Ήταν ένα πρώτο και αναγκαίο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά είναι ζωτική σημασία να αναπτύξουμε ένα υγιές και πλήρες μακροπροληπτικό πλαίσιο και για την Ένωση συνολικά και για τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση, αυτός ήταν στόχος προτεραιότητας του ESRB από τότε που δημιουργήθηκε. Πρώτα απ' όλα, για να υπάρξει μια ε, ε, στερεά βάση για προληπτικές ενέργειες κατά συστημικών κινδύνων, είναι ουσιώδες να αναπτύξουμε μακροπροληπτικές αρμοδιότητες και εργαλεία. Στην σύσταση που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, το ESRB τονίζει την ανάγκη για σωστό καθορισμό των μακροπροληπτικών αρμοδιοτήτων των εθνικών αργών για να μπορούν να δράσουν είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε ανταποκρινόμενες ε, στις συμβουλές του ESRB. Σύμφωνα με τα καθήκοντα του ESRB να παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεών του, οι πρώτες εκθέσεις από τα κράτη-μέλη που περιγράφουν τι πρόοδο έχουν ήδη σημειώσει θα πρέπει να ληφθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου με βάση το μηχανισμό συμμόρφωση ή παροχή εξηγήσεων του ESRB. Ένα βασικό δίδαγμα από το παρελθόν είναι ότι οι εντολέ για την οικονομική ή συστημική σταθερότητα πρέπει να συνοδεύονται από τη δυνατότητα και τα εργαλεία δράση. Οι μακροπροληπτικές αρχέ πρέπει να έχουν τον αναγκαίο εξοπλισμό μέσω αποτελεσματικών εργαλείων πολιτικής για να μπορούν να ανταποκριθούν με προληπτικό τρόπο στο πολύπλοκο και συνεχώ μεταβαλλόμενο περιβάλλον συστημικών κινδύνων. Το ESRB εργάζεται αυτή τη στιγμή για να καθορίσει τα ελάχιστα εργαλεία που είναι αναγκαία για να εφαρμόζονται μακροπροληπτικές πολιτικές παντού στην Ένωση. Δεύτερον, είναι ουσιώδες να διασφαλίσουμε ότι τα μακροπροληπτικά θέματα λαμβάνονται υπόψη όταν αναπτύσσεται, όταν εκπονείται η κοινοτική νομοθεσία για το χρηματοπιστωτικό τομέα, γιατί τα νομοθετήματα αυτά μπορεί να παίξουν ρόλο στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Υπάρχουν μια σειρά από σημαντικά ενωσιακά νομοθετήματα που παρακολουθεί το ESRB. Πρώτον, το σχέδιο οδηγίας και κανονισμού για ε, τα αναγκαία κεφάλαια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Είναι το λεγόμενο CRD-CRR. Δεύτερον, η πρόταση για να, υπάρξει, να υπάρξουν ρυθμίσεις για τα παράγωγα εκτός χρηματιστηρίου και, τα αποθετήρια ε, των συναλλαγών, το ΕΜΙΡ. Και δεύτερον, η πρόταση για την οδηγία Omnibus 2 που αφορά την επιτήρηση του ασφαλιστικού τομέα. Όσον αφορά το CRD-CRR, καλωσορίζω ιδιαίτερα την πρόσφατη πρόοδο που σημειώθηκε στην Επιτροπή σας, καθώς και στο Συμβούλιο, για να προωθηθούν οι προτάσεις που υπέβαλε η Κομισιόν πριν από λιγότερο από ένα χρόνο. Η εργασία σας μαζί με το Συμβούλιο αποτελεί πολλά υποσχόμενη βάση για να δημιουργηθεί ένα πολύ σημαντικό μακροπροληπτικό όργανο για να αντιμετωπιστούν οι συστημικοί κίνδυνοι των τραπεζών. Για να σας βοηθήσουμε και το Συμβούλιο για την εργασία σας στο crd το ESRB σας έγραψε το Μάρτιο, τονίζοντας μια σειρά από μακροπροληπτικών αρχών. Σας καλώ να λάβετε υπόψη τις αρχές αυτές, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι μακροπροληπτικές αρχές σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Είναι πλήρως εξοπλισμένες με ένα ευέλικτο σύνολο εργαλείων πολιτικής επαρκούς ε, πλαισίου που να τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν έγκαιρα την συσσόρευση συστημικών κινδύνων στο μέλλον. Φυσικά χρειάζεται επίσης σημαντικός ε, και αποτελεσματικός συντονισμός για να αποφύγουμε εξωτερικές ε, επιπτώσεις και παρενέργειες το ESRB είναι διατεθειμένο να παίξει κεντρικό ρόλο στην εργασία αυτή. Ήδη εργαζόμεθα για να δημιουργήσουμε ένα γενικό πλαίσιο για το συντονισμό των εθνικών μακροπροληπτικών πολιτικών από το ESRB εάν υπάρχουν διαμεθοριακές επιπτώσεις τέτοιων πολιτικών. Η συμφωνία για τον ΕΜΙΡ ήταν επίσης ε, σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την εφαρμογή των διδαγμάτων από την κρίση. Συμπεριλαμβάνει μια σειρά από χρήσιμα στοιχεία για να διασφαλίσουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ένωση. Το ESRB έχει ξεκινήσει την προπαρασκευαστική εργασία για να εκτελέσει τα καθήκοντα που του αποδίδει το ΕΜΙΡ. Από μάκρο προληπτική αντίληψη, ωστόσο, πρέπει να τονίσω ότι κατά τη γνώμη του ESRB το ΕΜΙΡ δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που τίθενται από την ενδεχόμενη προκυκλική επίπτωση της ε, διεύρυνσης ή προσπάθειας περιορισμού των ποιων ε, ε, προϊόντων θεωρούνται κατάλληλα για ε, εγγυήσει με βάση τις ευθύνες του. Το ESRB συνεχίζει να εξετάζει πώς θα μπορούσαν οι προϋποθέσεις της εγγύησης να χρησιμοποιηθούν ως μακροπολιτικό εργαλείο μεταγενέστερα. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ασφάλειες, για τον ασφαλιστικό τομέα, είναι σε φάση ε, εκπόνησης. Υπάρχουν σημαντικά ε, στοιχεία όσον αφορά για παράδειγμα τις εγγυήσεις, ε, τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις συζητιούνται αυτές τις μέρες και συμμετέχουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Το ESRB έχει υπόψη ότι διάφορα από τα θέματα αυτά έχουν ενδεχόμενα σχέση από μακροπροληπτική άποψη με την εργασία του ιδιαίτερα το νέο πλαίσιο Solvency 2, φερνικιότητα 2, μπορεί να διευρύνει την προκυκλικότητα των ισολογισμών των ε, ασφαλιστικών οργανισμών και ιδιαίτερα το επίπεδο των κεφαλαίων. Γι' αυτό, επειδή το αναγνωρίζουμε, σχεδιάζουμε διάφορα, πολιτικά, ε, διάφορα εργαλεία πολιτικής για να μετριάσουμε την προκυκλικότητα και άλλους παράγοντες. Είναι ζωτικό τα εργαλεία αυτά να σχεδιαστούν τόσο ώστε να δώσουν ένα σαφή και αξιόπιστο στόχο, ούτως ώστε η συνολική τους ε, δράση να έχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω μερικές μέσο πρόθεσμες διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που έχουμε υπόψη μας, που προσπαθούμε να αναπτύξουμε για να καταλάβουμε καλύτερα τις επιπτώσεις των συστημικών κινδύνων και για να εξακριβώσουμε με ποιους τρόπους μπορούμε να εργαστούμε για να έχουμε ένα πιο ανθεκτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ιδιαίτερα στρέφουμε την προσοχή μας στα διαρθρωτικά στοιχεία και του παραδοσιακού και του σκιώδου τραπεζικού τομέα. Πριν αναφερθώ στις εξελίξεις αυτών των τομέα, σε αυτούς του τομεί, να πω δύο λόγια για το συνολικό χρήμα, το πιστοτικό σύστημα που σε όλους τους τομείς του αυτή τη στιγμή μεταρρυθμίζεται. Σημαντικός στόχος αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι η διασφάλιση βιώσιμης παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από το σύστημα στην υπόλοιπη οικονομία. Στην Ευρώπη, ο χρηματοπιστωτικός τομέας ε, παραδοσιακά ε, βασιζόταν στις τράπεζες. Όμω μερικέ δραστηριότητε μπορεί να περάσουν σε άλλου τομεί όπου υπάρχουν λιγότερε ρυθμίσει. Στα προσεχή χρόνια. Ίσως ως άμεση επίπτωση της ε, πρόσφατης της τρέχουσας κρίσης και ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης των κανόνων για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τέτοιε εξελίξει μπορεί καταρχήν να ωφελήσουν το σύστημα αλλά πρέπει να επιτηρηθούν στενά για να περιοριστεί η δημιουργία νέων, ε, ε, νέων στοιχείων ε, ευάλωτων. Ας περάσουμε τώρα στον τραπεζικό τομέα. Η χρηματοπιστωτική χρήση μας απέδειξε ότι η, χρηματική, η χρηματοπιστωτική δομή των τραπεζών έχει προβλήματα και πρέπει να γίνει πιο βιώσιμη. ωστόσο, η δυνατότητα των τραπεζών να αντιμετωπίσει αυτές τις προσαρμογές δυσχεραίνεται από τις συνθήκες στον διατραπεζικό τομέα και τον μη ρυθμισμένο πιστοτικό τομέα. Οπότε χρειάστηκε όλο και περισσότερο οι τράπεζες να περάσουν σε καινοτόμα χρηματοδοτικά όργανα. Αναλύουμε αυτές τις αλλαγές των ε, συνθήκων χρηματοδότηση από μακροπροληπτική άποψη για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν παρενέργειες ή νέες συστημικές ε, ε, αδυναμίες. Η νεε συστημικες αδυναμιες η προσβαση σε περισσότερο ασφαλή χρηματοδότηση δημιουργεί βέβαια προβλήματα στο κεφάλι των τραπεζών. Αν πάει πολύ μακριά μια τέτοια πρόσβαση θα μπορούσε στο μέλλον να μειωθεί η σταθερότητα χρηματοδότηση ολόκληρου του συστήματος και με κυκλικό τρόπο να ενισχύσει την ε, έλλειψη πρόσβασης στις ιδιωτικές αγορές σήμερα. Επιπλέον, υπάρχουν ε, για παράδειγμα νέες καινοτόμες ε, μέθοδοι όπως οι ανταλλαγές ρευστότητας. Αυτά μπορούν να ε, μειώσουν το ή των τραπεζών. Ας περάσουμε τώρα στον σκιώδη τραπεζικό τομέα. Οι αστάθειες που προκύπτουν από ένα πολύ στενά αλληλεξαρτώμενο σύστημα καταδείχθηκαν από την οικονομική χρήση. Ο σκιώδης τραπεζικός τομέας ε, έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτήν την αλληλεξάρτηση, ιδιαίτερα λόγω των στενών σχέσεων μεταξύ του παραδοσιακού τραπεζικού τομέα και τον ε, περίπλοκο και μη διαφανή ε, παράλληλο τομέα. Έμεσα ή άμεσα βοήθησαν τα υψηλά επίπεδα αύξηση της μόχλευσης ορισμένες οικονομίες. Όπως γράφουμε στην ετήσια έκθεσή μας, το ESRB ήδη έχει αρχίσει να εργάζεται σε αυτό το τομέα. Χρειάστηκε, για παράδειγμα, να διαπιστώσουμε και να αποτιμήσουμε τους ενδεχόμενους συστημικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις νομισματικές αγορές στην τράπεζα και τα νομισματικά ταμεία και ε, σύμφωνα, ε, σύντομα θα δημοσιεύσουμε ένα ε, έγγραφο για αυτόν τον τομέα. Και είμαστε σε φάση εκπόνησης, το τελευταίο στάδιο εκπόνησης της συμβολής μας στην διαβούλευση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον σκυρόδη τραπεζικό τομέα. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους συστημικούς κινδύνους με βάση τους ε, ιδιαίτερους κινδύνους που προκύπτουν από τις διάφορες δραστηριότητες που υπάρχουν συνολικά στον σκιώδη τραπεζικό τομέα. Για παράδειγμα, πρέπει να εξετάσουμε την οικονομική φύση των ε, χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή, να δούμε τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν από τα προβλήματα και τις ανισότητες της ε, μόχλευσης και να δούμε σε τι βαθμό τα διάφορα ιδρύματα και οι διάφορες δοσοληψίες είναι ε, σωστά χρηματοδοτημένες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πλήρης μεταγραφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των, ε, πολιτικών, των πρωτοβουλειών πολιτικής που έχουν αποφαστεί σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερα αυτές που θα αναγγείλει το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στα πλαίσια αυτά το ESRB θα συνεργαστεί με όλους τους ενωσιακούς και διεθνείς θεσμούς και φορείς. Τονίζω λοιπόν ότι δραστηριότητε του SRB έχουν διεξαχθεί με την πλήρη συμμετοχή όλων των ε, θεσμών μελών του ESRB, ιδιαίτερα την ε, Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή, τη Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή και σε στενή συνεργασία με τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και προσβλέπουμε στην συνεχιζόμενη ε, επωφελή συνεργασία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, Μάριε. Είμαι βέβαιη ότι στις ερωτήσεις συνάδελφοι θα αναφερθούν σε, πρόσφατα, σε πρόσφατες εξελίξεις. Σχολίασε στην οδηγία για τις κεφαλαιακές ανάγκες και το Κοινοβούλιο πρέπει να τοποθετηθεί επ' αυτού και να αποφανθεί ας πούμε για πολλές λεπτομέρειες της οδηγίας αυτής Ιδίω για τις εγγυήσει και θέλουμε να μαζέψουμε όσε πληροφο... περισσότερες πληροφορίες μπορούμε για να καταλάβουμε καλύτερα τον σκιώδη τραπεζικό τομέα. Μία από τις διαστάσεις του βέβαια είναι πώς μπορεί να βλάψει τον επίσημο τραπεζικό τομέα και αυτό θέλουμε να το δούμε και στην ίδια την οδηγία για τον τραπεζικό τομέα. Γι' αυτό Αυτά συζητάμε στον τριμερή διάλογο. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα που θα τεθεί είναι από τον Πάμπλο Σάλμπα. Δύο-δύο τουλάχιστον να γίνονται οι ερωτήσεις για να οργανώσουμε καλύτερα το χρόνο μας. Ο Πάμπλο λοιπόν πρώτος και μετά η Μελίσσα. Ευχαριστώ για την παρουσίαση που μας κάνετε για πρώτη φορά την έκθεση της, ε, του ESRB μιλήσατε για, για ανασφάλεια μιλήσατε για αστάθεια αλλά όχι όσο τον προηγούμενο Νοέμβριο εγώ νομίζω ότι και τώρα είναι ασταθής η κατάσταση σοβαρή οι αγορές τιμωρούν με τρόπο άδικο και υπερβολικό χώρες που είναι απόλυτα φερέγγιες και που δρούν με υπεύθυνο τρόπο, λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις ε, τολμηρές. Γιατί για παράδειγμα να έχει ανέβει τόσο πολύ το επιτόκιο που πρέπει να πληρώσει η Ισπανία, ενώ προσπαθεί να εξηγιάνει τα φορολογικά η Ισπανία, προσπαθεί να μειώσει το έλλειμμα, προσπαθεί με αποφασιστικό τρόπο να κάνει διαθροτικές αλλαγές. Νομίζω ότι τα φορολογικά μέτρα που λήφθηκαν σε εθνικό επίπεδο, ενώ είναι τόσο σκληρές, δεν επαρκούν, δεν θεωρούνται επαρκείς από τις αγορές και δεν μας επιτρέπει αυτό να έχουμε πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Διερωτώ με, εάν μήπως αυτό που θέλουν να τιμωρήσουν οι αγορές είναι η έλλειψη αποφασιστικότητας και δράσης από την Ευρωζώνη συνολικά για να υποστηρίξει το νόμισμά του της και να υποστηρίξει ε, τα μέλη ε, της ε, Ευρωζώνης. Λέτε ότι, λέτε ότι αυξάνεται η αστάθεια. Πρέπει οπωσδήποτε στην ενέργεια της ε, Ευρωπαϊκής Τραγικής Τράπεζας να αποδώσουμε ευχαριστήσει γιατί κατάφερε να μειώσει το συστημικό κίνδυνο και να μειώσει την αστάθεια. Κύριε Ντράγκη, τι μπορεί να γίνει περισσότερο για να εγγυηθούμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τι συμπληρωματικά μέτρα συγκεκριμένα θα έπρεπε να υπάρξουν από τα χρηματοπιστωτικά θεσμικά όργανα της Ένωσης, ούτως ώστε να εγγυηθούμε την σταθερότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, Νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα γιατί έχουμε ακόμα 11 ερωτήσει ε, μέσα σε μισή ώρα. Πρέπει λοιπόν ε, να τι εξετάσουμε ανά τριάδα. λύς ε, και μετά Wolf. Έχετε δικαίωμα να μην απαντήσετε τίποτα, κανένα ερώτημα που να αφορά την Ευρωπαϊκή Τρική Τράπεζα. Ελίσσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξανά ήρθατε ενώπιόν μας. Θα ήθελα να μας πείτε ποιο είναι το κεντρικό στοιχείο της αντιμετώπισης του κινδύνου στην Ευρώπη. Εδώ ξέρουμε ότι υπάρχουν τα κρατικά χρέη, ότι παίζουν σημαντικό ρόλο οι τράπεζες, αλλά εξηγήστε μας λίγο Πώς τα διαχειρίζεστε αυτά, γιατί όλα γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα με την κρίση. Λοιπόν, πώς βλέπετε την αναδιοργάνωση ενός τέτοιου μηχανισμού αντιμετώπισης συστημικών κινδύνων. Τι εγγυήσεις προστασίας μπορούμε να έχουμε για τα τραπεζικά χρέη και τι εγγυήσεις για τα κρατικά χρέη. Ξέρουμε ποια είναι η εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά ειδικά ο σταθεροποιητικός μηχανισμός πώς θα λειτουργήσει, πώς θα καταλήξουμε σε αυτή τη μείωση του συστημικού κινδύνου. Δεύτερον, οι δικαιοδοσίες που έχουν προβλεφθεί για το ESRB, ποιες ακριβώς είναι ως προς την εποπτεία τουλάχιστον. Ο Βούλφ. Ευχαριστώ. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Καθήκοντα του ESRB είναι να αναλύει τους κινδύνους και να κάνει συστάσεις και προειδοποίησεις. Στην Ισπανία η ομάδα Μπάνκι έχει τεράστιες δυσχέρειες. Θα ήθελα να μάθω τι προειδοποίησεις και συστάσεις κάνατε προς την Μπάνκια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Δεύτερον, στην εφημερίδα Financial Times προτάθηκε ότι αν δεν μπορεί να υπάρξει φορολογική ένωση, να υπάρξει τουλάχιστον τραπεζική ένωση με ενιαίο σύστημα ασφάλισης και με ενιαία τραπεζική επιτήρηση. Ο Μπαρόζο υιοθέτησε αυτή την πρόταση. Θα ήθελα να μας πείτε αν νομίζετε κι εσείς ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να βοηθήσει να περιοριστούν οι συστημικοί κίνδυνοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όπως βλέπετε, θεωρούμε ότι είστε πηγή της γνώσης για όλα τα ζητήματα, παντός επιστητού. Ε, υπάρχουν ε, σκέψεις και για τους συστημικούς κινδύνους. Όσο μπορείτε, παρακαλώ δώστε μας μια απάντηση. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να απαντήσω και στα τρία ερωτήματα από κοινού. Όσο έναν βαθμό, Η απάντηση περιλαμβάνει τρία τμήματα που αφορούν ε, το κάθε ερώτημα. Τρία σημεία που αφορούν το κάθε ερώτημα. Αρχικά να σας πω ότι η χρηματοοικονομική κρίση που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, τέσσερα πλέον, έχει αλλάξει την αντίληψη που έχουμε για τον ε, κίνδυνο με ουσιώδη τρόπο και έχει αυξήσει την αποτροπή του κινδύνου ε, σε δραματικό βαθμό. Ξεκίνησε με το τραπεζικό σύστημα. Ε, τα ποσοστά μόχλευσης, τα οποία μέχρι τότε σε γενικές γραμμές θεωρούνταν αποδεκτά, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ξαφνικά. Έτσι είχαμε τον πρώτο γύρο ανακεφαλοποιήσεων, απομόχλευσης και το καθεξής. Μετά πήγαμε στα κράτη και τα ελλείμματα, τα εθνικά ελλείμματα. Επίπεδα ε, εθνικού χρέους ε, και ελλημάτων, τα οποία μέχρι τότε θεωρούνταν μακροπρόθεσμα βιώσιμα, πλέον θεωρούνταν μη βιώσιμα και μη διαχειρίσιμα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Και έτσι ο, ο χρονικός ορίζοντας ε, διαχείρισης ε, των προβλημάτων ξαφνικά γίνεται πολύ πιο σύντομος και έπρεπε, υπήρχε ανάγκη ανάληψης ε, δραστικών ενεργειών από τις κυβερνήσεις. Το ίδιο τώρα συμβαίνει και με την ε, σύνθεση της Ευρωζώνης. Ε, ένα σύστημα που είχαμε περίπου για 10 χρόνια, το οποίο θεωρούταν μέχρι τότε ε, βιώσιμο. Ίσως κατά μειοπικό τρόπο θα μπορούσα να πω. Τώρα φαίνεται ότι δεν είναι βιώσιμο, εκτός και αν αναλυφθούν άλλες ενέργειες. Αυτό ως προς το υπόβαθρο της τρέχουσας κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης πρέπει να, να ρωτηθούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μπορεί η Κεντρική Τράπεζα να καλύψει το κενό της ε, έλλειψης δράσης των εθνικών κυβερνήσεων ε, σε αυτό το τομέα. Και η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι ούτε το καθήκον μας, ούτε είναι αρμοδιότητά μας. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να καλύψει το κενό ε, δράσης στο, στο διορθωτικό τομέα από πλευράς κυβερνήσεων. Και πάλι όχι οι διαφορετικέ ε, μεταρρυθμίσεις, οι αναδιαρθρώσεις δεν έχουν σχέση με την ε, πολιτική επιτήρηση. Τέλος, μπορεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα να καλύψει το κενό της έλλειψης της ε, ε, διακυβέρνησης ε, της Ευρωζώνης και η απάντηση είναι και πάλι όχι. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Αυτό το, το είπα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προηγούμενη ακρόαση που είχαμε κάνει. Ουσιαστικά οι ηγέτες μας θα πρέπει να διευκρινίσουν το όραμά τους ε, για τα επόμενα χρόνια. Πώς, ποια θα είναι η υπόσταση του ευρώ μας στα επόμενα χρόνια. Ποιο είναι το ευρωπαϊκό όραμα που έχετε εσείς για τα επόμενα χρόνια. Όσο πιο γρήγορα το προσδιορίσουμε αυτό, τόσο το καλύτερο. Θυμάστε τον, ε, την, την πορεία μας για την ε, Νομισματική Ένωση. Το 1988 είχαμε, άνοιξε ο δρόμος και θέσαμε τους όρους που θα πρέπει να πληρούνται. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. να θέσουμε ένα τελικό στόχο και τους όρους που πρέπει να πληρούνται για αυτόν τον τελικό στόχο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό από πολλές απόψεις. Ε, σε πολλές κυβερνήσεις, σε περισσότερες χώρες, είναι σαν κάποιος ε, που προσπαθεί να διασχίσει ένα ποταμό, ε, αντιμετωπίζει πολύ ισχυρά ρεύματα και τώρα έχει φτάσει στη μέση. Εξακολουθεί να παλεύει αυτός ο άνθρωπος, αλλά ακόμα δεν βλέπει την άλλη όχθη, γιατί έχει ομίχλη. Εμείς σας ζητάμε αυτή τη στιγμή να διαλύσουμε αυτή την ομίχλη τα ρεύματα θα παραμείνουν ισχυρά και ο άναμος το ίδιο. Όμως θα βλέπουμε την τελική προοπτική. Αυτή είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά που μπορούν οι ηγέτες μας να κάνουν στην ανάπτυξη. Και αυτή η συμβολή θα μεταφραστεί σε μείωση ε, των, ε, των spreads και της ε, αποτροπής κινδύνου στο σύστημα. Και πάλι μια ιστορική αναδρομή. Θυμάστε ότι είχαμε αυτό τον, ε, την πορεία για την νομισματική ένωση και ξαφνικά το 1992 είχαμε το δανεικό ε, δημοψήφισμα που έθετε ένα αμφιβόλο αυτόν, ακριβώς, αυτή την πορεία προς την νομισματική ένωση και κατευθείαν τα επιτόκια αυξήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και έμειναν εκεί για πολλά χρόνια μέχρι που καταφέρουμε να ξεκαθαρίσουμε πάλι το τοπίο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα. Σε μια παρόμοια συγκυρία βρισκόμαστε. Και πρέπει να κάνουμε αυτά που σας πρότεινα προηγουμένω. Τώρα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό το όραμα. Μετά, πώς ε, θα λάβει η ουσιαστική μορφή αυτή η σαφήνεια του οράματος πρέπει, αυτό που είπατε ότι πρέπει να υπάρξει μια τραπεζική ένωση, δεν ξέρω αν αυτό είναι ο σωστός ε, όρο. Αυτό που προτείνεται ουσιαστικά είναι να, ε, να διαμορφώσουμε τρεις πυλώνες, ένα σχέδιο ε, ευρωπαϊκής ε, διασφάλισης ευρωπαϊκών καταθέσεων, Ταμείο Επίλυσης Κρίσεων και μεγαλύτερη κεντροποίηση της τραπεζικής επιτήρησης. Το Resolution Fund, αυτό το ταμείο, υποτίθεται ότι θα επιλύει, θα, θα χρηματοδοτεί την ε, την επίλυση κάποιων ε, τραπεζικών συστημάτων. Ουσιαστικά θέλουμε να, να, να διατηρήσουμε εν ζωή ε, σε όλα τα στοιχεία που είναι κρίσιμα για την λειτουργία του οικονομικού συστήματος, του τραπεζικού συστήματος, όπως τα, τα σχήματα πληρωμών. Ένας από τους στόχους λοιπόν θα ήταν αυτός. Αυτοί είναι οι τρεις ε, πυλώνες στους οποίους θα βασιστεί αυτό το σύστημα. Σε έναν βαθμό νομίζω ότι απαντώ σε πολλά από τα ερωτήματα που έχουν τεθεί, αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστώ. Θέλετε να συνεχίσετε επί του ιδίου θέματος. Όχι, για να καταλάβουμε. Όταν λέτε Ευρώπη εννοείται όλη την Ένωση ή την Ευρωζώνη. Μιλάμε για προβλήματα της νομισματικής ένωσης, του ευρώ. Δεν πρόκειται για προβλήματα ενωσιακά. Πρέπει όμως να σας θυμίσω ότι σε μια έκθεσή μας πριν από δύο χρόνια της Υγικής μας Επιτροπής είχαμε αναφέρει και με κάποιες λεπτομέρειες αυτά τα στοιχεία που ζητούσαμε να εφαρμοστούν και που προτείνετε κι εσείς πολλές φορές θα θέλαμε να είναι πιο συντονισμένες οι προσπάθειές μας με τις δικές αλλά τέλος πάντων επόμενα ερωτήματα Δόχια Σβέν και ο Ματίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Δέξια μετά την διάλυσή της ή μάλλον την εθνικοποίησή της περιόρισε πολύ τις δραστηριότητες της. Πέρυσι έφτασε το χρέος σε 11,6 δισεκατομμύρια και λένε ότι είναι κακή τράπεζα πλέον Πράγμα το οποίο πια έχει ήδη γίνει. Σύμφωνα με την Εθνική Βελγική Τράπεζα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η ανακεφαλαίωση της δέξια να γίνει πιο σύντομα από ό,τι αναμένουμε. Ενώ ερωτώ λοιπόν χρειάζεται η ανακεφαλαιοποίησή της. Και δεύτερον, η μέτοχή της δεν έδωσαν μόνο απαλλαγή στον πρώην πρόεδρό μας τον κύριο Σανλούκ Ντεάν αλλά του ζήτησαν και να μειώσει τα κεφάλαια κατά 4,1 δισεκατομμύρια πράγμα που άλλοι θεώρησαν σαν λογιστικό κόλπο για να αποφευθεί η ανακεφαλαιοποίηση. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Ο Σβέν. Ευχαριστώ Μάριε για την παρουσία σου εδώ. Είναι βέβαια σημαντικό και για μένα ως εισηγητή της δέσμης εποπτείας <clears throat> να ακούω τις πληροφορίες που μας έδωσες. Και εγώ είχα πολλές καλές εμπειρίες ως προς τη συνεργασία με το ESRB για νομοθετικά θέματα. Σε ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες που μας χορήγησες για θέματα όπως το Omnibus αλλά και τις δανειοδοτήσεις σε ξένο νόμισμα. Πρέπει όμως να πω ότι η αιτήσια αυτή έκθεση είναι κάπως μια χαμένη ευκαιρία γιατί εγώ θα ήθελα, ήλπιζα η έκθεση αυτή να δίνει ένα πλήρες όραμα, να κάνει μια πλήρη περιγραφή των μέσων επίτευξης της μακροοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής των κινδύνων ενώ τελικά είναι απλώς μια έκθεση πεπραγμένων. Δεν δίνει με αριθμούς ένα πλήρες όραμα, μια πλήρη περιγραφή του τι θέλετε να κάνετε. Δεν μπορείτε να το αλλάξετε και του χρόνου να έχετε μια πιο πλήρη περιγραφή και να κάνετε και μια ενδιάμεση έκθεση μεταξύ τώρα και του χρόνου. Και τώρα ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Το Δεκέμβριο πέρυσι υπόθηκε ότι θα χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση της Μπάνκια κατά 3 δισεκατομμύρια και τώρα μας λένε 19 ή 90. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Τι συστήνει το ESRB για να αποφύγουμε τέτοιου είδους διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις και για να είναι οι αριθμοί πιο αξιόπιστοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ντράγκη για την παρουσία σας. Ο συστημικός κίνδυνος είναι κάτι που δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε από άλλα προβλήματα. Θα χρειαστεί λοιπόν και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό να αναφερθώ και στις δραστηριότητες της ΕΚΤ γενικότερα. Η τωρινή κατάσταση στην Ευρωζώνη δείχνει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα χρηματοπιστωτικά μάλλον συστήματα, είναι αλληλένδετα σε, όλη την ευρωπαϊκή, σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Ίσως λοιπόν χρειαστεί βραχυπρόθεσμα κιόλας να γίνει μια αναδιάρθρωση των κρατικών χρεών. Μιλήσαμε για την Πάνκια γνωρίζουμε τα προβλήματα της Ισπανίας. Θα ανακεφαλαιοποιηθεί η μπάνκια λοιπόν. Μήπως έτσι αυξηθεί η πίεση των αγορών επί της χώρας αυτής και τότε θα αντιμετωπίσει η Ισπανία πραγματικά μια τραπεζική συστημική κρίση. Οι τράπεζες της Ευρωζώνης με το υπάρχον σύστημα ίσως συγχαίουν τα πράγματα στις δραστηριότητες τους. Ε, ρωτώ λοιπόν τα εξής. Πρώτον, κατά πόσον μπορούν οι τράπεζες στην κάθε χώρα να έχουν θετικά αποτελέσματα. Να είναι φερέγγιες. μήπως χρειαστεί ένα αποκεντρωτικό, αποκεντρωμένο σύστημα. Παρακαλώ να βιαστείτε γιατί λύγει ο χρόνος σας. Λοιπόν, αυτό που ρωτώ είναι το εξής. Είναι δυνατόν ή όχι. Να λυθεί το πρόβλημα από το κάθε κράτος χωριστά και πώς θα μπορούσε καλύτερα η Κεντρική Τράπεζα να ελέγξει το ενιαίο νόμισμα. Ευχαριστώ. Είχα πει ερωτήσεις και όχι λόγους. Να το θυμάστε όλοι. Μάριε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι σας συγχαίρω και εσάς προσωπικά και όλη την Επιτροπή. Το είχα πει και δύο χρόνια πριν. Νομίζω ότι μαζί είμαστε όλοι υπεύθυνοι και καλύτερα θα ήταν όντως όπως είπατε και εσείς να σας είχα ακούσει νωρίτερα τις προτάσεις σας. Για την ανακεφαλαιοποίηση της δέξια, αυτό είναι θέμα των εθνικών εποπτών, αλλά γενικότερα αυτό που δείχνουν οι περιπτώσεις της Μπάνκια και της Δέξια ε, ε, είναι ότι όποτε αντιμετωπίζουμε τις ζωτικές ανάγκες για ανακεφαλαιοποίηση πρέπει να σκεφτόμαστε την αντίδραση των μεμονωμένων εποπτών κυβερνήσεων που πάντοτε θεωρούν ότι υποτιμήθηκε η σημασία του προβλήματος και χρειάζεται λήψη επανειλημμένων μέτρων και πάντοτε των ίδιων και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Όλες οι χώρες αυτό έχουν κάνει. Αυτό όμως είναι ο χειρότερος δυνατός τρόπος αντιμετώπισης γιατί καταλήγουμε έτσι τελικά να κάνουμε το σωστό αλλά με το υψηλότερο δυνατό κόστος. Σας συστήνω λοιπόν όλους, όλες τις κυβερνήσεις να μην το ξεχνούν αυτό, ότι καλύτερο είναι να κάνει κανείς λάθος αντιδρώντας από την αρχή ίσως υπερβολικά παρά λίγο-λίγο και τμηματικά. Αυτό ισχύει και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Καλύτερο είναι να δούμε τα πράγματα ακόμη και υπερβολικά, με υπερβολική διαφάνεια, παρά να έχουμε ελλείψεις και να αναγκαζόμαστε να ξαναπάρουμε τα ίδια μέτρα. Το δεύτερο ερώτημα, πράγματι, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια ενδιάμεση έκθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Φυσικά γίνεται αυτό. Ο λόγος για τον οποίο η έκθεση αυτή προβλέφθηκε όπως προβλέφθηκε είναι γιατί βασίζεται σε ό,τι έκανε το ESRB μαζί με τους νομοθέτες. Είναι δηλαδή πολύ συγκεκριμένη έκθεση για συγκεκριμένα θέματα και δεν είναι μια γενική αξιολόγηση της κατάστασης. Αλλά μπορώ να δεχτώ την πρόταση σας αυτήν. Ευχαριστώ. Τώρα για την Πάνκια συγκεκριμένα. Και αυτό δείχνει αυτά που σας έλεγα πριν. Καλύτερο είναι να αντιδρούμε έστω και υπερβολικά αλλά από την αρχή παρά σιγά σιγά και τμηματικά. Χρειάζεται, αυτό δείχνει πόσο απαραίτητη είναι η κεντρική εποπτεία ιδιαίτερα για μεγάλους ομίλους που αντιμετωπίζουν και περισσότερο συστημικό κίνδυνο γιατί η Μπάνκια μπορεί να μην είναι διεθνής τράπεζα αλλά αντιμετωπίζει μεγάλο συστημικό κίνδυνο γιατί έχει μεγάλη συστημική σημασία. Τέλος, αν κατάλαβα καλά την τελευταία ερώτηση, ήταν τι θα μπορούσε να κάνει η ΕΚΤ για να διορθώσει κάπως να ελαφρύνει την κατάσταση στα χρηματοπιστωτικά. Κάναμε πολλά και πολύ γρήγορα. Ε, κόψαμε, μειώσαμε τα επιτόκια δύο φορές προβλέψαμε πιστώσεις σε δολάρια και και δύο φορές σας ανέφερα ήδη στην Επιτροπή σας τι κάναμε με τα LTRO. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις εγγυήσει ώστε να υπάρχει πρόσβαση και, για μεγάλες, και από μεγάλες αλλά και μικρομεσαίες τράπεζες, όλα αυτά έγιναν για να αποφύγουμε, για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι τράπεζες πέρυσι δηλαδή την έλλειψη κεφαλαίων, την έλλειψη χρηματοδότησης. Αρκεί αυτό για να ξαναρχίσουν οι τράπεζες να δίνουν δάνεια. Όχι. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι όπως η αποτροπή του κινδύνου. Έχουν βελτιωθεί βέβαια οι δανειοδοτήσεις από τον περασμένο μήνα, αλλά βασικά οι κεφαλαιακές ροές που παρατηρούμε, όχι σε όλες τις χώρες αλλά σε πολλές, είναι όπως είναι διότι υπάρχει μεγάλη αποτροπή κινδύνου ή φόβος του κινδύνου. Και η ΕΚΤ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Ο φόβος του κινδύνου συνδέεται με την έλλειψη χρημάτων αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα εμείς ως ΕΚΤ. Ευχαριστώ. Μεταξύ άλλων και γιατί είπατε ότι θα έπρεπε να ακούτε το κοινοβούλιο περισσότερο και νωρίτερα. Ίσως να το σκεφτεί αυτό και η Κομισιόν στους διάφορους τριμερείς διαλόγους που έχουμε μαζί τους και για το CRD και για το CRR. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω και αυτά που είπατε για τη διαφάνεια που είναι επίσης κάτι που θα μπορούσαν και οι χώρες μέλη να το λάβουν σοβαρότερα υπόψη τους. Η Μάρθα Αντρίσεν, Πολώνη και Μακάρθη. Η Μάρθα πρώτη. Ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση. Τι έννοια έχουν ε, τα τέσσερα αντοχής των τραπεζών που είχαμε πέρυσι για παράδειγμα και δεν βοήθησε να καθορίσουμε και να προλάβουμε περιπτώσεις όπως της Μπάνκια. Τι εκπλήξεις μπορούμε λοιπόν να αναμένουμε στο μέλλον. Δεύτερον, οι Ισπανικές τράπεζες ε, ε δυστυχώς πάσχουν από την φούσκα του κατασκευαστικού τομέα και χρειάζεται η Μπάνκια 19 δις. Οι τράπεζες αυτές έκαναν λανθασμένες αποφάσεις, όπως υπόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Πήραν λανθασμένες αποφάσεις. Γιατί να πληρώσουν για τις λανθασμένες ε, αποφάσεις του ιδιωτικού τομέα οι φορολογούμενοι. Η Ιρλανδία δεν είναι υπόδειγμα. Το ιδιωτικό χρέος μετατράπησε κρατικό χρέος και τώρα είναι στην εντατική Ιρλανδία. Ευχαριστώ. Ο Αλφρέντο. Πολώνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Ντράγκη. Οι πρόσφατες ε, χρηματοπιστωτικές αναταράξεις ε, κατέδειξαν την αναγκαιότητα να περιοριστεί η ε, αστάθεια των αγορών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τράπεζες. Βεβαίως η συμπεριφορά ε, των τραπεζών πρέπει να δευθωθεί, αλλά και των θεσμικών επενδυτών. Θεωρείτε ότι η μακροπροληπτική νομοθεσία είναι επαρκής για να εμποδίσει τους επενδυτές από το να πουλάνε υπερβολικά φτηνά τις μετοχές τους σε φάση αναταράξεων. Κάτι άλλο επίσης. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε για να ενθαρρύνουμε, να ενθαρρύνουμε συγγνώμη, ε, τους επενδυτές να κάνουν μέσο και μακροπρόθεσμες επενδύσεις και όχι ε, κινήσεις ε, σπασμωδικές. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν συμφωνείτε με διάφορους οικονομολόγους ότι ο μεγαλύτερος βράχυπρόθεσμος κίνδυνος για την σταθερότητα είναι το ότι αφαιρούν οι καταθέτες ε, τα χρήματά τους από τις τράπεζες τα στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα, 34 δις αφαιρέθηκαν από λογαριασμού στην Ελλάδα μέχρι το Μάρτιο 2012 και σε πολλές χώρες, ε, τις ε, χώρες είναι 3-2% λιγότερο, ενώ στη Γερμανία και τη Γαλλία ανέβηκαν κατά 6,5%. Ε, υποφελούνται και οι βρετανικέ τράπεζες. Τι εργαλεία λοιπόν θα μπορούσατε να δώσετε μέσω ενός πανευρωπαϊκού προγράμματος εγγύσεων, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκής ε, οι εγγύσεις αυτές. Τι προστασία μπορούμε να δώσουμε στους καταθέτες, τι εγγύσεις; Και αν ορισμένες ε, τράπεζες και ορισμένες χώρες δεν καλύπτονται, λόγω, για παράδειγμα, υποτιμήσεων, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι πολύ σωστό το ερώτημα. Εάν ένα, ε, έχουμε, αντιμετωπίσουμε συστημική κατάσταση των τραπεζών, τι μπορούμε να κάνουμε πρόεδρο. Ενδιαφέρουσε ερωτήσει κύριε δράγκη για να αντιμετωπίσετε. τα τεστ ε, αντοχής των τραπεζών θα τελειώσουν τον Ιούνιο του χρόνου ενώ τα προηγούμενα έγιναν ε, κατέληξαν πριν από περίπου ένα χρόνο. Αυτό καταδεικνύει άλλη μια φορά ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και οποιονδήποτε κεντρικών ε, μηχανισμών αποφασίσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή. Η περισσότερη συγκεντρωτικότητα της ε, εποπτείας των τραπεζών είναι αναγκαία, καταδεικνύεται και από την περίπτωση της Μπάνκια και άλλες. Απλούστερο νομίζω είναι να διαχειριστούμε κάποιες ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης εάν οι αποφάσεις παίρνονται σε πιο κεντρικό επίπεδο. Αυτό είναι νομίζω το δίδαγμα από τις εξελίξεις. Δεύτερη ερώτηση. Βεβαίως ε, και αυτή απόλυτα ορθή. Γιατί συνεχίζουμε να ξοδεύουμε χρήματα των φορολογουμένων για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Δηλαδή να καλύπτουμε τις τρύπε που ε, προκλήθηκαν λόγω αβάσιμων αποφάσεων του, του ιδιωτικού τομέα. Εξετάζοντας το μέλλον, ελπίζουμε η προληπτική νομοθεσία που σκοπεύουμε να ε, υιοθετήσουμε θα έχουμε δηλαδή ένα σύστημα επίλυσης που θα έχει δύο στόχους. Πρώτος θα είναι να μην χρησιμοποιούνται πλέον χρήματα των φορολογουμένων για να επιλύονται τα προβλήματα που προκύπτουν από συστημικούς κινδύνους. Και δεύτερον, να μην υπάρξει και πάλι αυτή η διακοπή στο σύστημα πληρωμών που προέκυψε μετά την κρίση της Λίμαν. Όλα όσα συζητήσαμε όλα όσα και εσείς ως Επιτροπή διερευνήσατε για πρώτη φορά πριν από δύο χρόνια, όντως αντιμετωπίζουν αυτά τα δύο θέματα. Προσβλέποντας λοιπόν στο μέλλον, νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτή η συνδυασμένη προσπάθεια και ε, συγκεντροποίηση της επιτήρησης και ένα σύστημα επιλύσεως των προβλημάτων που προκύπτουν σε τράπεζες. Αλλά τι συμβαίνει συχνά. Εάν κάποιες τράπεζες ε, πεθαίνουν μέσω ευθανασίας, ε, έχουμε ένα δίλημα. Είτε θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων, είτε ε, οι πιστωτές δεν θα λάβουν τα χρήματά τους. Θα προκύψει αφαιρεγκαιότητα. Και ξέρετε ότι αν δεν διαχειριστεί ένας φορέας με δυνατότητα επίλυσης της αφαιρεγγιότητας, τότε γίνεται συστημικό το πρόβλημα μεταδίδεται και μια τοπική τραπεζική κρίση γίνεται συστημική κρίση. Αυτό είναι πιστεύω ο κύριος λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις, όχι όλες βέβαια, κάποιες ε, τράπεζες ε, θανατώθηκαν. Αλλά είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει κάθε κυβέρνηση. Θα προκαλέσει συστημικό πρόβλημα ή όχι οποιαδήποτε απόφαση. Και αν θεωρούν ότι δεν θα προκαλέσει, οι κυβερνήσεις ε, κάνουν ευθανασία στις τράπεζες και βεβαίως ε, την πληρώνουν οι μέτοχοι αλλά και διάφοροι πιστωτές δεν ε, λαμβάνουν τα χρήματά τους. Είτε είναι εγγυημένα τα χρήματα αυτά ή όχι, εγγυημένε πιστώσεις ή όχι. Πώς να μειώσουμε την αστάθεια στον τομέα των κρατικών ομολόγων, ρωτήσατε επίσης. Κοιτάξτε. Να αναδιατυπώσω την ερώτηση. Πρέπει τα κρατικά ομόλογα να έχουν μη μηδενικούς ε, σταθμιστές κινδύνου. Μη μηδενική στάθμιση κινδύνου. Πρέπει το θέμα αυτό να το αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη σύνεση λόγω του θεσμικού πλαισίου που έχουμε στην Ευρωζώνη. Νομίζω ότι το ουσιώδες ερώτημα είναι τι προκάλεσε τέτοια υψηλή αστάθεια σε μια αγορά που ε, παραδοσιακά θεωρείται η ασφαλέστερη. Και παρερχόμεθα στους λόγους που προανέφερα. Είχαμε την φορολογική κρίση, είχαμε διαδροτική κρίση, είχαμε κρίση διακυβέρνησης. Οι τρεις αυτές κρίσεις δεν θεωρήθηκαν ζωτικής σημασίας, κρίσιμες, πριν τη χρηματοπιστωτική κρίση που τώρα έχουμε. Τώρα θεωρούνται. Αυτό έχει αυξήσει την αστάθεια σε όλες τις αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς κρατικών ομολόγων. Τελευταία ερώτηση, η απόσταση των καταθέσεων από τις τράπεζες που μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση. Μία απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να δανείζει της Φερέγγιες Τράπεζας. Θα συνεχίσει να διατηρεί ζωντανές και ενεργές τις γραμμές πίστοσης προς τις Φερέγγιες Τράπεζες. Και να σας ε, δώσω και ένα αποκλειστικό. Πριν από δύο-τρεις εβδομάδες αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε από τις δραστηριότητές μας χρηματοδότησης τέσσερις ελληνικές τράπεζες, διότι δεν πληρούσαν πλέον. Τα κριτήρια δεν ήταν επαρκής εταίροι στις ε, συναλλαγές αυτές μαζί μας, γιατί δεν είχαν επαρκές κεφάλαιο. Τώρα που υπήρξε η ανακεφαλαιοποίηση, αυτές οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες έγιναν και πάλι δεκτές στις ε, λειτουργίες ε, της νομισματικής πολιτικής. Η ΕΚΤΑΦ είναι λοιπόν διατεθειμένη να διατηρεί ζωντανές όλες τις γραμμές ρευστότητας προς τις φερέγγες τράπεζες. Υπήρξε και ένα ερώτημα για το μέγεθος αυτών των ταμείων. Ουσιαστικά από τις πλευράς των καταθετών ε, θέλω να σας ρωτήσω. Συνεχώς μιλάμε για το πώς θα σώσουμε τις τράπεζες, αλλά τι κάνουμε για τους ανθρώπους που ε, αποσύρουν τα χρήματά τους, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ε, να τα χάσουν λόγω υποτίμησης. Αν μιλάμε για έξοδο από την Ευρωζώνη, για παράδειγμα. Δεν θέλω να αφαιρθώ σε αυτό, λέει ο κύριος Δράγκη. Ναι, και κάποια από αυτά τα χρήματα πάνε εκτός Ευρωπαϊκής Ευρωζώνης. Θα αποφύγουμε την ε, ε, αυτό το φαινόμενο της, ε, της απόσυρσης των καταθέσεων όσο μπορούμε. Αν διαμορφώσουμε αυτό το, το Ταμείο Διασφάλισης των Καταθέσεων, αυτό θα ε, αποτρέψει την ε, μαζική απόσυρση, αλλά σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο. Δεν έχουν χάσει χρήματα οι καταθέτες λόγω ε, πτώχευσης τραπεζών μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Γιατί μιλάμε για την κατάσταση πριν από δύο χρόνια. Πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον. Συμφωνώ απολύτω από αυτού, λέει ο κύριος Δράγη. Εντάξει, συνεχίζονται οι συζητήσεις. Έχουμε δύο ακόμα ερωτήσεις και θα φτάσουμε πιο γρήγορα στην ψηφοφορία αν κάνετε ησυχία. Επομένω παρακαλώ όσοι έχουν φτιάξει πηγαδάκια να σταματήσουν. Σόφι Ιντερβέλ και Γιάνγκο Φέλ. Σόφι. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Θα επαναλάβω ένα ερώτημα που σας είχα υποβάλει κατά τη διάρκεια του ε, διαλόγου εποπτεία και είπατε ότι μπορώ να σας απαντήσω μόνο όταν, ε, φορώ, όταν έχω με, την ιδιότητα του διευθυντή του ESRB. Αυτό κάνω λοιπόν και εγώ εδώ τώρα. Πώς αξιολογείτε ε, το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους στο Ολλανδικό σύστημα στεγαστικών δανείων. Και δεύτερον, έχετε αξιόπιστες και, πλήρης, ε, και επαρκείς πληροφορίες για το συντεξιδιωτικό σύστημα και για τράπεζες που ενδεχομένως να έχουν συστημικό αντίκτυπο στην Ευρώπη και βρίσκονται εκτός Ευρώπης. Thank you. Please, can I... Παρακαλώ να σταματήσουν οι επιμέρους συζητήσεις γιατί δεν θα συνεχίσουμε σε αντίθετη περίπτωση. Παρακαλώ σταματήστε. I'll start naming and shaming if you keep on Θα αρχίσω να σας ε... κατονομάζω αν συνεχίσετε έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ, Sharon. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ντράγκη. Και να θέσω δύο ερωτήματα άμεσα. Πρώτον, ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Την 1η Ιουλίου ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα τεθεί σε ισχύ. Υπάρχουν αντικρουόμενες ε, απόψεις ε, για το κατά πόσο μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα κονδύλια τράπεζες ε, για την ανακεφαλοποίησή τους. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θα μπορούν οι τράπεζε να αξιοποιήσουν αυτά τα κονδύλια, αυτό το ταμείο για την ανακεφαλοποίησή του. Δεύτερον, το δεύτερο ερώτημα συνδέεται με τον συστημικό κίνδυνο. Θα ήθελα να μου πείτε αν προβλέπετε κάποιο μηχανισμό, αν για παράδειγμα ε, έχουμε το, το φαινόμενο της μαζικής απόσυρσης από τους καταθέτες, γιατί είναι σημαντικό ο τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να χρηματοδοτεί την οικονομία. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, η Εθνική Κεντρική Τράπεζα των Κάτω Χωρών έχει ε, ε, αποστείλει προειδοποιήσεις για αυτό το ζήτημα. Λέει ότι ανησυχεί ιδιαιτέρως. Θα δούμε ποια βήματα προτείνουν και θα τα συζητήσουμε στο ESRB στην επόμενη Ολομέλεια, σίγουρα τον Ιούνιο. Ενδεχομένως και πριν από αυτό, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε αναλάβει δράση λοιπόν επ' αυτού. για το δεύτερο ερώτημα. Οι περισσότεροι από εμά ε, το έχουμε αυτό κατά νου μετά την εμπειρία με το EFSF. Πώ είμαστε σίγουροι ότι θα, ε, θα λειτουργήσει καλά το ESM. Ε, μπορεί να έχουμε πολλά χρήματα, αλλά να μην μπορούμε να τα αγγίξουμε. Είναι σαν να μην τα έχουμε ουσιαστικά για πολλούς λόγους, ε, εν μέρη λόγω και της ε, κακής εμπειρίας ε, στο παρελθόν, εγώ δεν είμαι σίγουρος για το κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί ο ESM. Ακόμα και τώρα οι εμπειρογνώμονες ε, προσπαθούν να βρουν τρόπους ε, για την αξιοποίηση του ESM για την ανακεφαλοποίηση τραπεζών. Το θέμα βέβαια δεν είναι αν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά αν μπορεί να γίνει άμεσα, ε, χωρίς να περάσουμε από, την, περάσουμε από τις κυβερνήσεις. Γιατί εάν αποδεχθούν να έχουν ένα μνημόνιο κατανόηση με το ESM, με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα, τότε μπορούν να το αξιοποιήσουν για την ανακεφαλοποίηση τραπεζών. Είναι όμω μια σκέψη που έχουμε κατά νου, δεν θέλουμε να επαναληφθεί ε, το φαινόμενο του παρελθόντος και νομίζουμε ότι με το ESM, ε, με τον μηχανισμό στήριξη, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος, ρωτήστε για τους ε, καταθέτες που μπορούν να αποσύρουν τις καταθέσεις τους. Το ίδιο ερώτημα με προηγουμένως κατ' ουσίαν. Ε, φοβόμαστε ότι θα υπάρξει μια τέτοια, ένα τέτοιο φαινόμενο. Ε, η απάντηση είναι ότι μπορούμε, έχουμε τα απαραίτητα μέσα για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο ε, σε ό,τι αφορά τις αφαιρέγγιες τράπεζες. Κάτι ρωτήσατε για τα στεγαστικά σωστά. Είπατε για τα, για τα ασφαλιστικά ταμεία, στεγαστικά ταμεία. Είπα, αν έχετε τις απαραίτητες και επαρκείς πληροφορίες και για τις τράπεζες εκτός Ευρώπης. Ε, ο ESRB θεωρείται μηχανισμός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για την Ευρωζώνη. Είπα και προηγουμένω ότι η μεγαλύτερη συγκεντρωποίηση τη εποπτεία είναι ένα απαραίτητο στοιχείο, αλλά αναφερόμουν ε, στι ε, τράπεζε τη Ευρωζώνη. Γι' αυτό απάντησα εν μέρη στην ερώτησή σα. Τώρα, για να έχουμε πληροφορίε για τι τράπεζε εκτό τη Ευρωζώνη, αλλά εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αναφέρεστε σε αυτές, τότε έχουμε πληροφορίες. Για τις υπόλοιπε τράπεζε εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτές λοιπόν λαμβάνουμε κάποιες πληροφορίες μέσω της συνεργασία μας με άλλες εθνικές εποπτικές αρχές. Ε, ε δεν βρίσκεται στο πεδίο δραστηριοτήτων ε, της ε, ESRB. Παρ' όλα αυτά, εμείς ε, είμαστε αρκετά φιλόδοξοι και γι' αυτό έχουμε έρθει σε επαφή, έχουμε συνεργασία με άλλους φορείς. Παρ' όλα αυτά θέλουμε περισσότερα. Θέλουμε να έχουμε πραγματική, ειλικρινή ε, ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του ESRB. Αυτό έλεγα και προηγουμένω. Ιδίω ό,τι αφορά την Ευρωζώνη, μπορούν πολλά ακόμα να γίνουν για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Ευχαριστώ. Σας κατευχαριστώ γιατί απαντήσατε σε τόσες πολλές ερωτήσεις. Τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία, θα προεδρεύσει η Νταρλίν. Σας αφήνω λίγα λεπτά για να αναπαυτείτε.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 and uh, so this was again stupid, so we, we had a basic agreement but not fixable. That's, the report of the semester. Yeah. What I would like to know if, um, colleagues, take, take your seats for... Παρακαλώ καθίστε, λάβατε θέσεις. Είπα να τα κάνουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα με τη συνεργασία σας μπορούμε να το πετύχουμε. Can I και όσοι θέλουν να φύγουν να κάνουν τις ιδιωτικές τους συζητήσεις εκτός αιθούσης, διότι έχουμε καθυστερήσει κατά 10 ολόκληρα λεπτά. Λοιπόν, δοκιμή με τις κάρτες σας. Δοκιμή. Παρακαλώ ψηφίστε πλασματικά. Όσοι δεν είχαν βρει το σθένος να πατήσουν το κουμπί παρακαλώ να το πράξουν γιατί δεν το πάτησαν όλοι. Εγώ θα έχω την κάρτα μου σε δύο λεπτά. Καλά θα περιμένουμε μετά όταν έρθει να μας πείτε. Μου τη φέρνουν από το γραφείο μου. Α, ωραία. 34, ακόμα 4 λείπουνε. Όχι εσάς, σας ε, σημείωσα εσάς, σας σημείωσα. Θα σας τη φέρω από το γραφείο. Λοιπόν. Ωραία. Λέω τώρα να γίνουν πρώτα με το χέρι οι ψηφοφορίες εκτός αν υπάρχει πρόβλημα. Τότε θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Λοιπόν, αρχίζουμε με την έκθεση Κράτσα για την ελκυστικότητα των παιδιών 40, τροπολογία 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 που είναι συμβατή υπέρ. Κατά. Όχι. Θα επαληθεύσουμε, θα επαληθεύσουμε. Έχω τους αριθμούς όμως, παρακαλώ να προσέχετε. Για τη 42 ηλεκτρονική. Έληξε. 17 υπέρ 22 κατά. Απορρίπτεται. Το πρωτότυπο κείμενο ή όχι, όχι, όχι. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ. Συμβιβαστική β υπέρ. Κατά ε, ε, ε, εγκρίνεται και αυτή. Συμβιβαστική γ. Α, είναι γλωσσική, εντάξει, καλά, γλωσσική είναι. Γα, είπαμε συμβιβαστική Γ υπέρ, εγκρίνεται. 53, υπέρ. Εγκρίνεται 54 υπέρ. Εγκρίνεται συμβιβαστική δέλτα. Εγκρίνεται 57 υπέρ. Εγκρίνεται 58 υπέρ. Εγκρίνεται προφορική τροποποίηση 59 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται νομίζω. Να την επαληθεύσω την 59. Να την επαληθεύσω. Την επαληθεύω. Εγκρίνεται, εγκρίνεται, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Όχι την 59 λοιπόν, 60 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ. Εγκρίνεται. Α, κατά τμήματα. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα της συμβιβαστικής ε. Λοιπόν, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 66 υπέρ απορρίπτεται 67 υπέρ όχι θα το επαληθεύσουμε θα το επαληθεύσουμε το 67 δεν είναι 67 67 έληξε 15 υπέρ 24 κατά απορρίπτεται Χρειάζεται να ψηφίσουμε το πρωτότυπο. Όχι, όχι, όχι. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, το πρωτότυπο υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική Φεφ. υπέρ. Α, είναι πάλι κατά τμήματα. μέχρι εκεί το πρώτο τμήμα, μέχρι εκεί που λέει τόσο μαζικά στο μέλλον υπέρ Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Περιότι και τα λοιπά. Υπέρ. Κατά. Και αυτό εγκρίνεται. Συμβιβαστική ζήτα. G. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Επαλήθευση. Απορρίπτεται σαφώς. 76 υπέρ. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 78 υπέρ. Εγκρίνεται. Παράγραφος 17 το πρωτότυπο κείμενο υπέρ. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Απορρίπτεται το πρωτότυπο κείμενο τη 17, 18 μάλλον, ε, υπέρ, εγκρίνεται, 80 και 81 ταυτόσημες. Υπέρ, υπέρ, εγκρίνεται, 82 υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τα H υπέρ, εγκρίνεται. 86 υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική I θ υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική J. Για δύο τμήματα, σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα χωρίς τη φράση που αναφέρει εδώ. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, μόνον αυτή η φράση, ναι, υπέρ, εγκρίνεται και αυτό. Από ό,τι βλέπω, γιατί ο κύριος ομάδες είναι υπέρ, λοιπόν. 93 υπέρ. Εγκρίνεται 94 υπέρ. Εγκρίνεται 95 υπέρ. Εγκρίνεται 96. Εγκρίνεται 97. Εγκρίνεται 98. Εγκρίνεται 99. 99. Επαλήθευση. Έληξε 17 υπέρ 24 ε, κατά. Απορρίπτεται. Το πρωτότυπο κείμενο υπέρ. Εγκρίνεται το σκεπτικό τώρα. Μπορούμε να το πάρουμε όλα μαζί το 1 μέχρι 8 ή όχι. 1 με 8 μαζί. Α, πρέπει πρώτα την 100, την 100 υπέρ. Την 100. Δεν είχαμε ψηφίσει την 100. Οι ελεύθεροι τι λένε, υπέρ ή κατά. Κατά, τότε απορρίπτεται. απορρίπτεται. απορρίπτεται. Το πρωτότυπο κείμενο υπέρ. Εγκρίνεται. Τώρα τα σκεπτικά 1 με 8. Ναι, λοιπόν, 1 με 8. Υπέρ εγκρίνονται. Το πρωτότυπο για το 33 με 34 εγκρίνεται επίση. Τροπολογία 9, κ. Γκίγκολ, Ντιπέρ. Νομίζω ότι απορρίφθηκε θα επαληθεύσουμε. Απορρίφθηκε. Έχουμε μια προφορική τροπολογία, τη 10 υπέρ, εγκρίνεται. 11 υπέρ, εγκρίνεται. Το πρωτότυπο κείμενο υπέρ, εγκρίνεται. 12 υπέρ, εγκρίνεται. 13 με προφορική τροποποίηση Δεν ψηφίσαμε το πρωτότυπο, το ψηφίσαμε, το ψηφίσαμε. Εγώ είμαι πιο γρήγορη από εσά. Λοιπόν, 13 έχει αποσυρθεί. Σβέν την απέσυρε. λοιπόν. Το πρωτότυπο. Το πρωτότυπο. Υπέρ. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Εγκρίνεται. 16 υπέρ εγκρίνεται 17 εγκρίνεται 18 εγκρίνεται 19 έχει καταπέσει το πρωτότυπο κείμενο όχι 20 20 περ εγκρίνεται 21 εγκρίνεται 22 εγκρίνεται 23 εγκρίν, ε, υπέρ 23 υπέρ απορρίπτεται 24 υπέρ απορρίπτεται 25 υπέρ απορρίπτεται 26 υπέρ εγκρίνεται 27 υπέρ εγκρίνεται 28 υπέρ εγκρίνεται 29 με προφορική τροποποίηση την έχετε λοιπόν. εγκρίνεται 30 υπέρ εγκρίνεται 31 εγκρίνεται 32 εγκρίνεται 33 εγκρίνεται J, το πρωτότυπο κείμενο δηλαδή. 33 υπέρ, εγκρίνεται. Το πρωτότυπο του λάμδα υπέρ, εγκρίνεται. 34 υπέρ, εγκρίνεται. Για το σκεπτικό νη, συμβιβαστική J, α υπέρ, εγκρίνεται. 38 υπέρ, εγκρίνεται. 39 υπέρ εγκρίνεται. Μετά οι γνωμοδοτήσεις, μία μόνο χρειάζεται να ψηφίσουμε, τη Ήτρε. Παρακαλώ υπέρ. Επαλήθευση. «25 υπέρ 16 κατά» εγκρίνεται. 4 της Ήτρε υπέρ κατά εγκρίνεται 4 της Ήτρε 4 της Ήτρε επαλήθευση μάλιστα επαλήθευση Ήτρε 4 12 υπέρ 27 κατά απορρίφθηκε Ήτρε 8 υπέρ εγκρίνεται τα άλλα καλύπτονται από τις συμβιβαστικές. Παράγραφος 14, τροπολογία 14 σε δύο τμήματα της Ήτρε. Πρώτο τμήμα μέχρι το μικρό σίγμα υπέρ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, το υπόλοιπο, απορρίπτεται. Τώρα πολλές τροπολογίες της Ήτρε, μία-μία. 15 της Ήτρε υπέρ. Εγκρίνεται 16 υπέρ. Απορριπτέται 17 της Ήτρε υπέρ. Εγκρίνεται 18. Εγκρίνεται 19. Εγκρίνεται. Και μετά από την περιφερειακή τροπολογία 1 υπέρ. Εγκρίνεται 2 περίφ απορρίπτεται Τρία περίφ εγκρίνεται θέλετε επαλήθευση για την τρία. θα την επαληθεύσουμε θα την επαληθεύσουμε Τρία. έληξε 19 υπέρ 22 κατά απορρίπτηκε τέσσερα της περίφ υπέρ Εγκρίνεται. 7 της περι... 7 της Περιφερειακής Επιτροπής. Εγκρίνεται και αυτή. 11 της Περιφερειακής υπέρ. Εγκρίνεται 13 της Περιφερειακής με προφορική τροποποίηση. Εγκρίνεται και αυτή. 14 της Περιφερειακής. Απορρίπτεται. 16 της περιφερειακής. Α, απορρίπτεται. 17 της περιφερειακής. Απορρίπτεται. Όχι. Μα αν είσαστε υπέρ τότε θα έχει εγκριθεί. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. εντάξει. Λοιπόν, 17 υπέρ. Εγκρίνεται. 18 με προφορική τροποποίηση υπέρ εγκρίνεται και η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικός για το κείμενο όσο έχει τροποποιηθεί άρχεται η ψηφοφορία εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ και 3 κατά και 4 αποχές συγχαρητήρια τι έχουμε τώρα Okay. So we now are moving. Να περάσουμε τώρα. Στην έκθεση της κυρίας Κόκονη. Yes, yes, yes, you can correct me. Okay. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Συμβαστική α υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική β υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική γ εγκρίνεται. Συμβαστική δ υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. 15 τροπολογία 15 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ. 75 Ωραία. Απορρίπτεται. Συμβαστική ε υπέρ. Τροπολογία 82 υπέρ. Απορρίπτεται. Αλλά θα το ελέγξουμε νομίζω. 82 παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος. Απορρίπτεται. 22 με 19 ήταν όντως ε, μικρή διαφορά. Συμβαστική F υπέρ. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. 97. Απορρίπτεται. Αλλά παρόλα αυτά να το ελέγξουμε παρακαλώ. Νομίζω ότι είναι ίδια η... ο ίδιος ο σχετισμός, αλλά για να ελέγξουμε. Ωραία. Πέρας. 18-23. Όχι ακριβώς, όχι ακριβώς ίδιος σχετισμός. Συμβαστική G υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ. Τροπολογία 20 υπέρ. Εγκρίνεται. Συγγνώμη. Να ελέγξουμε το H. Ωραία. Να ελέγξουμε. Αλλά νομίζω ότι εγκρίθηκε. Αλλά ας ελέγξουμε. Εντάξει. Πέρασε. 31 με 9. Εγκρίνεται σαφώς. Ωραία. 20 υπέρ. Εγκρίνεται. 107 υπέρ. Απορρίπτεται. 110 υπέρ. Λοιπόν, 111 δεν χρειάζεται προηγούμενη υπέρ. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Εγκρίνεται. Δεν χρειάζεται προηγούμενη γιατί λόγω της ε, προηγούμενης ψηφοφορίας. 10 από τη νομική υπέρ. Εγκρίνεται. Καλός έλεγχος. Νομίζω ότι απορρίπτεται γιατί είδα ότι άλλαζε η σηματοδότηση από τους ε, συντονιστές. Αλλά ας το ελέγξουμε. Κύριε Πρόεδρε, σας συγχαίρω για το πόσο γρήγορα πηγαίνετε. Αλλά οι διερμηνείς δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τόσο σύντομα. Και καμιά φορά χανόμαστε. Ναι, βεβαίως κερδίζουμε χρόνο, αλλά, αλλά να... Μα νομίζω ότι όλοι έχετε το κατάλογο ψηφοφοριών, λέει η Πρόεδρος αλλά ακόμη και οι συντονιστέ τα χάνουν, λέει ο κύριο Γκοζέ. Δέκα λοιπόν, νομική. 17-23. 17 υπέρ, 23 κατά. Απορρίπτεται. 11. Ωραία, απορρίπτεται. Συμβαστική I. Υπέρ. Εγκρίνεται. 1-1-8. Υπέρ. Απορρίπτεται. Γιατί βλέπω ότι καταψηφίζουν δύο μεγάλες ομάδες. Συμβαστική J υπέρ. Α, με συγχωρείτε. Η τροπολογία 9. Ε, συγγνώμη, 119 υπέρ. Η συμβαστική J υπέρ εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εγκρίνεται, εγκρίνεται, σαφέστατα. 121 υπέρ. Εγκρίνεται. Ωραία, σε ελέγξουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δύο δεν ψήφισαν ακόμη, παρακαλώ ψηφίστε πριν κλείσει η ψηφοφορία. Ωραία, πέρας. 16 υπέρ 23 κατά, 24 κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική κάπα υπέρ εγκρίνεται. 123 εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ εγκρίνεται. 16 έμπλ υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική M εγκρίνεται. Τροπολογία 131 υπέρ. Επίσης εγκρίνεται. N υπέρ. Συμβαστική εγκρίνεται. 34 υπέρ εγκρίνεται. Να περάσουμε στα 135 υπέρ. Α, καταπίπτει γιατί εγκρίναμε την 34. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε την 137. Τροπολογία 35 υπέρ. Πρέπει να το ελέγξουμε. Γιατί νομίζω ότι 35 λοιπόν. Όχι απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Τροπολογία ε, γνωμοδότηση 1 υπέρ της απασχόλησης υπέρ. Τροπολογία 36 κλούτερς υπέρ απορρίπτεται. Τροπολογία 1 οκονή εγκρίνεται. Πάμε στην αιτιολογική ΙΑ υπέρ. Ε, 1α συγγνώμη. Εγκρίναμε την 71 γιατί τότε δεν χρειάζεται. Ωραία, ας ψηφίσουμε. 37 λοιπόν. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Επίσης εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Απορρίπτεται. 47 υπέρ απορρίπτεται 48 υπέρ εγκρίνεται 1 νομική υπέρ απορρίπτεται 4 υπέρ εγκρίνεται 49 α δεν χρειάζεται α όχι χρειάζεται χρειάζεται α, α μάλιστα καταπίπτει τροπολογία 3 έμπλ υπέρ εγκρίνεται αλλά να το ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 κατά 21 υπέρ. Τροπολογία 51 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Εγκρίνεται. 4 έμπλε Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Εγκρίνεται. Ωραία. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική παρακαλώ. Άρχεται για το κείμενο το νομοθετικού, του νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται. Πέρας. 35 υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. ...36 υπέρ, μάλιστα, και ο κύριος Κλίντς. Για, για το νομοθετικό ψήφισμα, λέει η πρόεδρος. Για το νομοθετικό ψήφισμα άρχεται. Εντάξει. Πέρας. 37 υπέρ και δύο εποχές σε καθευτηρία. We're Ας ψηφίσουμε τώρα. Αν θέλετε καθίστε παρακαλώ. Ψηφίζουμε για την 70 υπέρ. Υιοθετείτε. Συμβαστική α υπέρ. Υιοθετείτε. Μετά 74 υπέρ. Συγκρίνεται 75

Uh, I can also check how many people are voting at the same time, and only 36 people are. 36 άτομα ψήφισαν. Μένουν ακόμα δύο. Είκοσι υπέρ, 17 κατά. Υιοθετείτε. Συμβαστική Β, υπέρ. Υιοθετείτε. Συμβαστική Γ, υπέρ. Υιοθετείτε. Συμβαστική Δέλτα υπέρ. Υιοθετείτε. Τροπολογία 97. Υπέρ. Υιοθετείτε. 98. Υπέρ. Υιοθετείτε. Συμβαστική Ε. Υπέρ. Υιοθετείτε. Συμβαστική F. Υιοθετείτε. 110. Ε, Απορρίπτεται, αλλά θα το επαληθεύσουμε. Παρακαλώ. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, 27 κατά. Συμβαστική G. Α, πρέπει να κάνω την 111 υπέρ. Φιλελεύθερη. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω, στο ελέγξουμε. Uh, Απορρίπτεται. Συμβαστική G υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 130 υπέρ. Απορρίπτεται. 131 εγκρίνεται. 132. 133 εγκρίνεται. 17 απορρίπτεται 18 υπέρ απορρίπτεται 19 υπέρ απορρίπτεται η συμβαστική Α υπέρ εγκρίνεται 138 υπέρ εγκρίνεται 121 138 θέλετε να ελέγξω Ωραία, ελέγχουμε τη συμβαστική I. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 30-12 δεν ήταν τόσο μικρή διαφορά, αλλά θέλετε τα λέμε. 138 υπέρ. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΙ Εγκρίνεται. Τώρα να δούμε την 24 υπέρ του εισηγητή 25 υπέρ. Α, είστε κατά τώρα. Τότε απορρίπτεται. Ωραία. 25. 25 παρακαλώ. Είστε κατά. Απορρίπτεται. 26. 26. Ωραία. Απορρίπτεται και αυτή. Συμβαστική IB εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ εγκρίνεται. 28 υπέρ εγκρίνεται. 29 υπέρ. 30 υπέρ. Ίδια με 146. 31 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική J. A θα ελέγξω. Αλλά μόνο μία ομάδα καταψηφίζει. Αλλά αφού θέλετε, εντάξει. Για την 31 λοιπόν έλεγχος. Εγκρίνεται. 23 με 20. Μηδέν αποχέ. Συμβαστική J, α, υπέρ. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις, 36, υπέρ. Εγκρίνεται. 35 υπέρ εγκρίνεται. 37 υπέρ εγκρίνεται. Νομική 1 υπέρ εγκρίνεται. 38 εγκρίνεται. 39 εγκρίνεται. Ξέρω, αλλά μόνο μία ομάδα καταψηφίζει. Εγώ από ψηλά βλέπω καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ελέγξουμε. Νομίζω ότι είναι ίδιος ο συσχετισμός. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι είναι ίδιος. Α, δεν ήταν μεγάλη διαφορά, 21-20. Απορρίπτε για την 21-21 τελικά. Είναι η ψήφος του κυρίου Κλίντς. Κύριε Κλίντς, έχετε κάρτα. 38 απορρίπτεται, 39 υπέρ. είναι κατά. Είστε εσείς υπέρ. Εγκρίνεται τότε. Η 39. 40 υπέρ. Να ελέγξουμε τη 39. Ωραία. Πέρας. Απορρίπτεται. 21 υπέρ, 22 κατά. Τροπολογία 40 υπέρ. Πρέπει να τις ελέγξουμε όλες αυτές. Λοιπόν, ελέγχουμε την 40. «25-15 περνάει. 41 υπέρ. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Εγκρίνεται. 44. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Εγκρίνεται. Μα Βίκυ θες να ελέγξω αλλά η ομάδα σου είναι υπέρ. Ε, τροπολογία 1 του εισηγητή εγκρίνεται. Συμβαστική κάπα υπέρ εγκρίνεται. 51 υπέρ εγκρίνεται. 53 υπέρ απορρίπτεται. Σαφώς. Συμβαστική L υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 59 εγκρίνεται. Αλλά παρόλα αυτά θα ελέγξουμε. 59 δεν είναι απόλυτα σαφές. Πέρας. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Εγκρίνεται. 6 υπέρ με τα 65 οπότε γίνεται και αυτή 7 οι 7 και 67 ίδιες είναι μια μιας απάλληψης ε, υπέρ εγκρίνεται 68 υπέρ 8 υπέρ εγκρίνεται 9 υπέρ εγκρίνεται 10, 10 υπέρ εγκρίνεται Ωραία να την ελέγξουμε τη 10. 21 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται. 69 εγκρίνεται. Δύο τελικές ψηφοφορίε ηλεκτρονικές. Πρώτη για το τροποποιηθέν κείμενο. Πέρας. 33 υπέρ, 3 κατά, 4 αποχές. Και τώρα να ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα ηλεκτρονικά. Α, πριν ή μετά τη ψηφοφορία. Νομίζω ότι ήδη έγινε και η δεύτερη ψηφοφορία. Δεν ψήφισαν ακόμη όλοι, περιμένατε. 34 υπέρ, 2 κατά. 35 υπέρ, 2 κατά, 3 αποχές. Και τώρα η Σοφή και εγώ θα θέλαμε να μας δώσει εντολή η Επιτροπή να αρχίσουμε τη διαγραμματεύση με το Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι δημιουργεί πρόβλημα, αλλά όπως ξέρετε η Δανέζικη Προεδρία εξέφρασε σοβαρή επιθυμία να κλείσει αυτό το θέμα. Συμφωνείτε κυρία Οκονή. Απολύτως, λέει η κυρία Οκονή, όπως και ο Φίλιπ Λαμπέρ. Και εγώ θα ήθελα να ψηφίσουμε να υπάρξει διαπραγματευτική εντολή για το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Ωραία. Συμφωνούμε, καλούμε την ε, Επιτροπή, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον εισηγητή και του Σκιώδης, να αρχίσουν διαπραγματεύσει. Κλείσαμε το θέμα αυτό. Ο πρώτος τριάλογος θα γίνει, τριμερής διάλογος, θα γίνει 4 Ιουνίου, κοινό ε, τριμερής διάλογος με το Ταμείο αυτό της κοινωνική επιχειρηματικότητα. Θα συμμετάσχει και αυτό δηλαδή στον τριμερή διάλογο. Okay, Λοιπόν, η επόμενη ψηφοφορία. Έκθεση Κλούτα. Πρόσβαση σε βασικές ε, θεμελιώδεις ε, τραπεζικές υπηρεσίες. Συμβαστική Α, υπέρ. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 73, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο, λοιπόν, υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 82 υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική Δ υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική Ε υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ εγκρίνεται εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ επίσης εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική N υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική π υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική R ε, εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική ταφ υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική U υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική V υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική W υπέρ εγκρίνεται. Θα μας τελειώσει το αλφάβητο σε λίγο. Τροπολογία 195 γκουλάρ υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική X υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 200 υπέρ. Απορρίπτεται. Το αρχικό λοιπόν κείμενο υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική Y εγκρίνεται. Συμβαστική Z εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΑ εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΒ εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΣ εγκρίνεται. Συμβαστική, ε, συγγνώμη, τροπολογία 219 υπέρ. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική AD εγκρίνεται. Συμβαστική AE εγκρίνεται. Και μετά το αρχικό κείμενο, αιτιολογικέ σκέψει 1 προ 10, αιτιολογικέ αναφορέ 1 προ 10 εγκρίνονται. Τροπολογία του κυρίου Κλούτε επίση εγκρίνεται. Συμβαστική AF εγκρίνεται. Συμβαστική AG εγκρίνεται. Συμβαστική AH εγκρίνεται. Τροπολογία 14 εγκρίνεται. Συμβαστική AI εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 18 και 19 που είναι ταυτόσιμες για απάλληψη υπέρ εγκρίνεται οπότε δεν ψηφίζουμε το πρωτότυπο τροπολογία 20 υπέρ εγκρίνεται συμβαστική AJ εγκρίνεται συμβαστική AK εγκρίνεται τροπολογία 26 ποιοι είναι υπέρ απορρίπτεται Ωραία, ας ελέγξουμε την 26. Σαφώς απορρίπτεται. Τροπολογία AL υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική AM υπέρ. AN υπέρ εγκρίνεται. AO εγκρίνεται. AP εγκρίνεται. AR εγκρίνεται. Τώρα να ψηφίσουμε την 55. Απόρριπτεται. Πρέπει... AS υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ εγκρίνεται. 61 υπέρ εγκρίνεται. 62 υπέρ εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το τροποποιηθέν κείμενο άρχεται. Πέρας. 36 υπέρ, 37 υπέρ, 2 κατά, 0 αποχές, χαρακτήρα. Μακάρι να ήταν όλες τι ψηφοφορίε έτσι. Και να καταλήγαμε σε καλούς ε, συμβιβασμού. Καλά τα πάμε. Είναι 11 παρα 5 και έχουμε ακόμα 2. Τώρα να δούμε το την έκθεση του κυρίου Σκυκλούνα, 20 κύριοι λόγια ανησυχία των επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη λειτουργία τη ενιαία αγορά. Συμβαστική Α υπέρ εγκρίνεται. Μετά 3 υπέρ εγκρίνεται. 5 υπέρ. Απορρίπτεται νομίζω. Α το ελέγξουμε γιατί κάποιοι έχουν φύγει. Ελέγχουμε λοιπόν την 5. Πέρας ψηφορίας. 17 υπέρ, 22 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ, εγκρίνεται. 6 υπέρ, εγκρίνεται. 7 υπέρ. Ε, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Believes towards unemployment and poverty. Υπέρ. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Stress, solidarity and democracy. Και αυτό απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Και πάλι σε τμήματα. Το is concerned μέχρι basic foodstuffs. Απορρίπτεται. Μετά το δεύτερο, τρίτη πρόταση υπέρ. Υιοθετείται, σαφώς. 13. Απορρίπτεται. Συμβαστική γάμα υπέρ. Υιοθετείται. Παράγραφος 4 του αρχικού κειμένου υπέρ εγκρίνεται, 16 υπέρ εγκρίνεται, 17 υπέρ εγκρίνεται, 18 υπέρ εγκρίνεται, 19 εγκρίνεται, 23 υπέρ εγκρίνεται, 20 έχουμε προφορική τροπολογία αλλά την έχετε μπροστά σας υπέρ εγκρίνεται, 21 υπέρ Τη φιλελεύθερη. Απορρίπτεται τότε. 22 υπέρ. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Εγκρίνεται. 26. Εγκρίνεται. 27. Εγκρίνεται, στο επαληθεύσουμε όμως. 27. Για την 27. 27, 27. The vote is open on 27. Um, it Εγκρίνεται 21 με 19. 28 υπέρ. Εγκρίνεται 29 υπέρ. Εγκρίνεται 30 υπέρ. Εγκρίνεται 31. Προφορική τροπολογία υπέρ. Εγκρίνεται 32 υπέρ εγκρίνεται. 33 υπέρ με προφορική τροπολογία εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορία. And the vote is closed. Πέρας. 35 υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Σε χαρητήρια στον κύριο Σικλούνα. Hey. Okay. Okay. So, now we're Ωραία. Τώρα, του κυρίου Λαμπέρ για πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ε, για την ανάκληση τη 1364, δηλαδή Ευρωπαϊκέ Ενεργειακέ Υποδομέ για κατάργηση τη απόφαση. Πρώτη τροπολογία του εισηγητή, υπέρ ε, εγκρίνεται 45 υπέρ εγκρίνεται, 46 ε, υπέρ εγκρίνεται, 47 υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική Α με ψηφορία κατά τμήματα. Τρει μάλιστα τέτοιε ψηφορίε. Πρώτο τμήμα, where appropriate energy infrastructure categories, υπέρ απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, projects involving at least κτλ. Υπέρ. Υιοθετείται. Να το ελέγξουμε. Το ήξερα θέλετε να το ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Υιοθετείτε 22 υπέρ, 17 κατά. Τρίτο τμήμα, που είναι το υπόλοιπο υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Υιοθετείτε. 61 υπέρ. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Εγκρίνεται. 63 καταπίπτει. 10 υπέρ. Εγκρίνεται. 64. Απορρίπτεται. 65. Απορρίπτεται. 66. Εγκρίνεται. 67. Εγκρίνεται. 11. Απορρίπτεται, νομίζω. Ας το ελέγξουμε. Ναι, απορρίπτεται 17 υπέρ, 21 κατά. 68 υπέρ. Ναι, ναι, ναι. Απορρίπτεται. σχεδόν όλοι είναι κατά, αλλά αν θέλετε στο ελέγξουμε, εντάξει. Α, 19 προς 18, άρα υιοθετείτε. Μάλιστα, 12 υπέρ. Υιοθετείτε. 13 υπέρ. Εγκρίνεται 69 υπέρ. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. 15 παρακαλώ. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Ας την ελέγξουμε. 21 υπέρ 17 κατά, εγκρίνεται 16 υπέρ, εγκρίνεται 71 υπέρ, απορρίπτεται 72 υπέρ, εγκρίνεται νομίζω, ναι, ξεκάθαρα, δεν κοιτάζουμε το 17, 18 υπέρ, εγκρίνεται, Ναι. Εγκρίνεται. 20 υπέρ, 18 κατά. 73 υπέρ. 73. Απορρίπτεται. 74 υπέρ. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. 20. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Απορρίπτεται. 21 υπέρ τη ηγητή. Το ίδιο νομίζω ισχύει και εδώ, αλλά στο ελέγξουμε για την 21. Πέρας. 17 υπέρ, 21 κατά. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Εγκρίνεται 86 υπέρ. Εγκρίνεται 22 υπέρ. Εγκρίνεται 23 υπέρ. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Και αυτή εγκρίνεται. 88 υπέρ. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Και αυτή απορρίπτεται. 90 υπέρ. Απορρίπτεται. 91 υπέρ. Για την 91 θέλουμε πρώτα. Εγκρίνεται. 92. Αλλά είπατε να τα δείτε από κοινού. Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. 92 υπέρ. Εγκρίνεται. 93 υπέρ εγκρίνεται. 24 υπέρ, εγκρίνεται. 25 υπέρ, εγκρίνεται. 26 εγκρίνεται. 94 απορρίπτεται. 95 υπέρ. Ας την ελέγξουμε την 95. 19 με 18 εγκρίνεται λοιπόν. 96 υπέρ. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Απορρίπτεται. 100 εγκρίνεται. 101 υπέρ. Εγκρίνεται και αυτή. 27 υπέρ. Απορρίπτεται, άρα την ελέγχουμε όμως. 18 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. 28 υπέρ. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Απορρίπτεται. 29 και 30 ε, αποσύρθηκαν. 31 υπέρ. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Απορρίπτεται. Μετά πάμε στις ιδεολογικές σκέψεις. 33 υπέρ. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Το ελέγχουμε. 25 με 13. 34 υπέρ. 34 εγκρίνεται. 35 υπέρ. Ελέγχουμε το 35. Έναρξη ψηφοφορίας. ...21 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. 37 υπέρ. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Εγκρίνεται 40. Απορρίτεται. 41. Εγκρίνεται 42. Εγκρίνεται 43. Εγκρίνεται 44. Εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, πριν ε, κάνετε την τελευταία ψηφοφορία, Νομίζω ότι μόνο εκ μέρου του ονόματό μου θέλω να σα ευχαριστήσω για την αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα με την οποία κάνατε αυτή τη ψηφοφορία. Ναι, ίσω ήμουν πολύ γρήγορη. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν, αλλά αν το έχετε μπροστά σα, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε και πρόβλημα, γιατί δεν ήθελα να τελειώσουμε μετά τι 11. Τα... Το πετύχαμε. Νομίζω ότι λίγη ψηφοφορία για το τροποποιημένο κείμενο έναρξη ψηφοφορία. And the result is 36 υπέρ 0 κατά και 2 μόνο αποχές. Και για το ε, νομοθετικό ψήφισμα έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας, 34 επέρ, 0 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε your Uh, και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας στην ψηφοφορία και συγγνώμη που έτρεχα λίγο. In the end we got there. Thank you. Nothing to announce. Ευχαριστώ. Next point on the agenda, which is the last one. Okay. Well, let's some clear. We, I'm going to... Because I was... Right. Uh, <coughs> Επόμενο θέμα είναι το 18. Το σύστημα φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών διαφορετικών κρατών μελών, παρένθεση αναδιατύπωση. Κλείνει η παρένθεση. Η κυρία Πέλτς είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σύντομα, πολύ σύντομα μάλιστα, θα σας περιγράψω το γιατί χρειάζεται διαφοροποίηση, αναδιατύπωση του συστήματος. Καταρχήν υποστήριζω την πρόταση της Κομισιόν για τις τροποποιήσεις που χρειάζονται για να επιτευχθεί ο στόχος της μεταρρύθμισης του συστήματος. Τον Σεπτέμβριο του 2011 είχαμε εγκρίνει την νέα μορφή της οδηγίας PEN και την CCTB και τον Απρίλιο φέτος το Κοινοβούλιο κατέληξε ότι πρέπει να αυξηθεί η φορολογική συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών για κάποια εναρμόνιση. Επίσης τέθηκε το θέμα της φοροδιαφυγής που δημιουργεί τεράστια απώλεια εσόδων ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που γνωρίζουμε σήμερα με τα ελλείμματα και τα χρέη. Ο στόχος είναι να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή και την μη φορολόγηση, είτε είναι εθελοντική είτε όχι, σκεμμένα είτε όχι. Έτσι ώστε να καταλήξουμε στην αντικατάσταση των ισχυών των κανόνων για εξαιρέσεις και να μειωθούν ή, ή να επανεξεταστούν οι μειώσεις των φόρων που χορηγούνται σε διάφορα ιδρύματα. Γενικά συμφωνώ με τις προτάσεις της Κομισιόν, αλλά θα ήθελα επίσης να τονίσω το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αναθεώρηση αυτή της οδηγίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Πέλτς. Με χαρά θα διαπιστώσατε ότι είμαι σε θέση να μιλήσω μαλτέζικα. Ο κύριος Βάνοκ είναι παρόν. Α, με συγχωρείτε. Δεν ήξερα ότι είστε σκιώδης. Λοιπόν, Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κομισιόν προτείνει αναθεώρηση της οδηγίας 2349. Καλό είναι αυτό, γιατί πράγματι δεν μπορέσαμε να καταργήσουμε όλους τους φραγμούς στην εσωτερική αγορά, ιδιαίτερα για τις δημοθεωριακές πληρωμές. Η ύπαρξη των συστημάτων φορολόγησης ήδη από την καταβολή του μισθού θέλει να αποφύγει τη διπλή φορολόγηση. Η Κομισιόν προτείνει το, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας να διευρυνθεί και να συμπληρωθεί ο κατάλογος των οντοτήτων που έχουν δικαίωμα σε μειώσεις φόρων. Εφόσον βέβαια ο φόρος πληρώνεται πράγματι στο κράτος προέλευσης. Πολύ καλή η προσέγγιση αυτή Πρέπει όμως να διασφαλιστεί ότι το κείμενο της Κομισιόν δεν θα δίνει καμία δυνατότητα για φοροδιαφυγή. Και οι τροπολογίες της κυρίας Γκάλ Πέλτς είναι σωστές. Εκτός από αυτό, από την αποφυγή δηλαδή της διπλής φορολόγησης, πολύ σημαντικό θα ήταν επίσης να διασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργήσουμε δεύτερη μη φορολόγηση που να καταλήγει τελικά σε πλήρη φορολογική απαλλαγή. Γι' αυτό καταθέσαμε τροπολογίες και χαίρομαι εκ των προτέρων για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να συνεννοηθούμε με την κυρία εισηγήτρια και τους υπολείπους σκιώδης. Ευχαριστώ. Τώρα ο Σβέν, εξ ονόματος των Πρασίνων. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά μου θυμίζουν την οδηγία μητρός θυγατρός. Έχουμε ήδη ξανασυζητήσει παρόμοια θέματα και με τους ίδιους συναδέλφους. Δυστυχώς δεν έχουμε πλήρης δικαιοδοσία συναπόφασης. Αν είχαμε θα άλλαζαν τα πράγματα. Την περασμένη φορά είχαμε πολύ στεναρή θέση και παίξαμε πολύ σημαντικότερο ρόλο γιατί το Συμβούλιο δεν ήταν και ενθουσιασμένο με όλα όσα ζητούσαμε. Τώρα όμως χαιρόμαστε που συζητιέται το θέμα αυτό και τη γενική κατεύθυνση των προτάσεων της Κομισιόν Επίσης θεωρούμε ότι η έκθεση της ηγητρίας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλώς θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει κάποια συνέπεια μεταξύ αποφάσεων που ήδη έχουμε λάβει και της τωρινής έκθεσης. Δηλαδή πρώτον θεωρούμε ότι θα ήταν καλό να προσθεθεί μια γενική ρήτρα αντισύγχυσης που ζητούσαμε ήδη από τον Απρίλιο σε ψήφισμά μας για τη φοροδιαφυγή. Αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στη χρήσιμη σας έκθεση και επί τα δεύτερον δηλαδή να υπάρξει μεγαλύτερη συνέπεια με την απόφασή μας για την οδηγία μητρός και θυγατρός. Να υπάρχει δηλαδή ένα ελάχιστο ποσοστό φορολόγησης. Αυτό νομίζουμε ότι χρειάζεται γιατί βλέπουμε ότι στο Συμβούλιο η παλαιότερη συζήτηση ξαναγίνεται και μερικές χώρες μέλη θέλουν να ενθαρρύνουν την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων χαμηλής φορολόγησης υπονομεύοντας έτσι τη συνέπεια του φορολογικού καθεστώτος που ισχύει σε διάφορες χώρες. Η συνήθιση ύποπτη στο Συμβούλιο τα λένε αυτά, η Ιρλανδία, Αγγλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο. Πάντα τα ίδια γίνονται, αλλά αφού έχουμε ενιαίο νόμισμα πρέπει να έχουμε κοινού κανόνες, αλλιώς πρέπει να πάψουμε να ζητάμε κοινή φορολογική και οικονομική πολιτική, γιατί θα καθιστούμε ακόμη πιο δύσκολη την νομοθεσία που θα ισχύει σε όλες τις χώρες. Εδώ το Κοινοβούλιο νομίζουμε ότι πρέπει να συνεχίσει την ίδια κατεύθυνση που είχε πάρει και προηγουμένως και υποστηρίζουμε την εισηγήτρια στις βασικές της ιδέες. Θα καταθέσουμε μερικές υποστηρικτικές τροπολογίες για να αυξηθεί η συνέπεια με προηγούμενες αποφάσεις. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ρεαλίστριες. Θα ανταγωνιστούμε το Συμβούλιο, αλλά υπάρχει απέτηση της ομοφωνίας. Και επομένως το θέμα είναι αν θα υπάρξει όχι ενισχυμένη συνεργασία. Αν όχι, τότε θα χρειαστεί να περιμείνουμε μέχρι τη συντέλεια του κόσμου για να ληφθούν αυστηρά και αποφασιστικά μέτρα αποφυγής της φοροδιαφυγής που δεν θα τα καταλάβουν και κανένας συμπολίτης μας, ούτε συμπολίτρια. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον ομιλητή των συντηρητικών. Ίσως ε, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για τις ενδιαφέρουσες και πολύτιμες προτάσεις τους. Ε, στον Σβέν θα μπορούσα να πω ότι προσπαθώ να ευθυγραμμίσω την έκθεση αυτή με την προηγούμενη οδηγία για το CCTV. Ελπίζουμε να υπάρξει σημαντική και ισχυρή πλειοψηφία και εδώ και στην Ολομέλεια. Ωραία. Η προθεσμία για την ε, για την υποβολή τροπολογιών είναι η 7η Ιουνίου. Η Επιτροπή θα ψηφίσει στις 9 Ιουλίου και ε, θα πάει στην Ολομέλεια η έκθεση